Welcome, uh, Καλώς ήρθατε συνάδελφοι, ευχαριστώ που ήρθατε για την συνεδρίαση. Όπως βλέπετε δεν είμαστε όλοι εδώ, αλλά έχουν έρθει αρκετοί. Πρώτο θέμα λοιπόν είναι η έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Όχι. Α, Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεδομένης της σημερινής απόφασης από το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας, εμείς δεν έχουμε λάβει ακόμα κάποια απόφαση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επαναλαμβάνει ότι έχει 751 ναι, ευρωβουλευτές, 748 έχουμε στην πραγματικότητα. Το θέμα της ε, ασυλίας των τριών καταλανών ευρωβουλευτών είναι θέμα αρμοδιότητός μας. Οπότε θεωρώ ότι μετά από τρεις μήνες ε, που έχει συσταθεί το Κοινοβούλιο θα πρέπει επιτέλους να ληφθεί μια απόφαση για την ασυλία αυτών των τριών. Προτείνω λοιπόν να τεθεί στην αριστερή διάταξη. Τουλάχιστον να γίνει μια συζήτηση για το θέμα. Μάλιστα. Έγινε αυτή η πρόταση. Ε, υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους δεν είναι καλή ιδέα αλλά η απλούστερη απάντηση είναι να ψηφίσουμε. Όποιος θέλει λοιπόν να συζητήσουμε το θέμα της Καταλωνίας μπορεί να μας πει. Όσοι δεν είναι υπέρ, παρακαλώ πείτε μου. Ωραία. Ε, σαφώς απορρίπτεται, οπότε δεν θα μπει στην σημερινή ημερήσια διάταξη άλλα σχόλια για τη σημερινή ημερήσια διάταξη. Ωραία. Οπότε εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Σημείο 2 είναι το ότι ο κύριος Λαγκοντίνσκι, ο οποίος απουσιάζει, ζήτησε η VDR, η γερμανική τηλεόραση, να μας κινηματογραφήσει. Θα ήθελαν να πάρουν κάποια πλάνα από την αρχή της συνεδρίασης για να παιχτούν στην εκπομπή Europa Magazine. Έχετε κάποια αντίρρηση, όχι ευχαριστώ. Οπότε μπορείτε να συνεχίσετε. 2β. Ανακοινώσεις της Προέδρου αποφάσεις των συντονιστών. Στις 26 Σεπτεμβρίου 2019 οι συντονιστές έλαβαν τις εξής αποφάσεις. Αποφάσισαν για την ε, κατανομή των εκθέσεων για την απαλλαγή του 2018. Για το δικαστήριο θα είναι ο κύριος Ζιλ Λεμπρετόν. Αποφάσισαν η γραμματεία να πάει ως παρατηρητής ε, στις ε, συναντήσεις του διαλόγου των συμμετεχόντων του άρθρου 17 της οδηγίας για το copyright στην ενία ψηφιακή αγορά και ορίστηκε ο Τίμο Βόλκον ως ε, εκπρόσωπος της Επιτροπής μας στη, στο πάνελ ΣΤΟΑ. Σημείο 3. Ανταλλαγή απόψεων με τον ε, εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Καλωσορίζω τον κύριο Αρσαμπό, εκτελεστικό διευθυντή, ο οποίος θα μας παρουσιάσει το σχέδιο πολιτικού στρατηγικού προγράμματος για τα επόμενα πέντε χρόνια. Έτσι το Κοινοβούλιο θα μπορέσει να εκφραστεί για την στρατηγική αυτή. Κύριε Αρσάμπο, λοιπόν, σας ευχαριστώ που ήρθατε και σας δίνω τον λόγο. Thank you, Madam Chair. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Δικαστικών Νομικών Υποθέσεων, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ πολύ που θα έχουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων για, το, για την κατεύθυνση που θα πάρει το Γραφείο Πνευματικής Διοκτησίας, όπως ε, προβλέπεται σχετική νομοθεσία. Ξέρετε ότι είναι αποτέλεσμα συνεργασία ε, με την Ευρωπαϊκή Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα με την Επιτροπή Γιούρη. Θέλουμε να ενισχύσουμε αυτή τη σχέση. Για να σα μιλήσω για το επόμενο στρατηγικό σχέδιο, θα ήθελα να αναφερθώ πρώτα ε, στο γιατί το EUIPO αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε όπως εξελίχθηκε η μεγαλύτερη δηλαδή υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ξεκινάμε ε, το, το Αλικάντε πριν από 25 χρόνια το 1994 όταν δημιουργήθηκαν τα γραφεία μας αλλά Πρώτα διαπιστώσαμε ότι πρέπει να κάνουμε κάτι έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα προστατεύσουμε τα πνευματικά δικαιώματα για να εξασφαλίσουμε την ευημερία των πολιτών και των επιχειρήσεων. Θέλησαμε πρώτα να έχουμε ευρωπαϊκά τέτοια δικαιώματα με το ευρωπαϊκό σήμα. Ο νομοθέτη όμω είχε πάντα κατά νου ότι πρέπει να υπάρχει μια υπηρεσία με ευρύτερε αρμοδιότητε στον τομέα των πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτό οδήγησε σε μια εξέλιξη ε, του πεδίου δραστηριοτήτων τη ε, υπηρεσία μα ε, με το, τη δημιουργία του, ε, μεταξύ άλλων το 2012 του, ε, του, Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την παραβίαση αυτών των πνευματικών δικαιωμάτων. Μεταξύ άλλων η υπηρεσία μας ε, με τη νέα την ονομασία EU IPO περιλαμβάνει ε, συνεργασία για ζητήματα μεταξύ ιδιοκτησίας εκτός, εντός, εντός μάλλον και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ αρμοδιοτήτων των απαιτήτων μας. Αυτό αποτυπώνει ότι e, το EUIPO IPO πλέον συνεισφέρει σχεδόν σε όλους τους τομείς ε, πνευματικών δικαιωμάτων και βεβαίως πέρα από τα σήματα ε, και τα διπλώματα βελτιστεχνίας στα ευρωπαϊκά εξακολουθεί να είναι αυτό ένα σημαντικό στοιχείο των μας, είναι αυτό που ε, εγγυάται και την ανεξαρτησία την οικονομική μας. Δύο εκατομμύρια ε, αιτήματα είχαμε για τα πληρώματα ε, για, μάλλον για σήμα κατά τεθέν, και αυτό είναι που δείχνει πόσο δημοφιλείς είμαστε. Θα πρέπει επίσης να λάβατε το τελευταίο, τελευταία έκθεση για τις παραβάσεις στον τομέα των μαρικών δεξιών όλε τι έρευνε που έχουμε κάνει, είναι ενδιαφέρον ε, το ενδιαφέρουσα έκθεση αυτή να τη διαβάσετε και δείχνει και ποιε είναι οι προτεραιότητε τη ε, υπηρεσία μου για τα επόμενα πέντε χρόνια. Δεν θα επαναλάβω όλα τα αριθμητικά στοιχεία. Είναι πάνω από 40 οι έρευνε που έλαβαν χώρα. Αλλά κάποια αριθμητικά στοιχεία νομίζω αξίζουν τον κόπο, αξίζει τον κόπο να τα αναφέρω. Οι επιχειρήσει που χρησιμοποιούν πνευματικά ε, δικαιώματα ε, design, διπλώματα ευρεσιτεχνία, ε, αλλά και γραφικέ ενδείξει, είναι υπεύθυνα για ένα σημαντικό ποσοστό ε, τη απασχόληση και τη ανάπτυξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια πρόσφατη μελέτη τη υπηρεσία μα και τη υπηρεσία πατεντών δείχνει ότι τα τελευταία τρία χρόνια η συνεισφορά στο ΑΕΠ αυτών των επιχειρήσεων έχει αυξηθεί στο 45%, κατά 45%, 6,6 τρισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, ο αριθμό των θέσεων εργασία που άμεσα ή έμεσα προέρχονται από αυτέ τι επιχειρήσει έχει αυξηθεί κατά 39%. 96% ε, των εξαγωγών τη Ευρωπαϊκή Ένωση επίση αφορά τι επιχειρήσει αυτέ. Ε, Πολλέ μελέτε δείχνουν ότι τα, τα πνευματικά δικαιώματα χρησιμοποιούνται με διαφορετικού τρόπου. Θα δούμε στην έκθεση ότι αυτέ οι εταιρείε είναι πιο ανταγωνιστικέ, παράγουν ε, θέσει εργασία ε, καλύτερη ποιότητα, μεγαλύτερη ποιότητα και πιο καλοπληρωμένε. Πρέπει όμω να υπάρξει ένα πιο καλό συντονισμό με τα εθνικά συστήματα πνευματική ιδιοκτησία και με τι αρχέ επιβολή τη νομοθεσία αυτή κυρίω. Σύγκριση, ε, σύγκριση, σύγκληση, μάλλον ε, σύμπραξη είναι πολύ σημαντικά στοιχεία για να εξασφαλίσουμε ότι οι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει θα έχουν την υποστήριξη που χρειάζονται, έτσι ώστε να κεφαλοποιήσουν την δημιουργικότητά του, την καινοτομία του και να δημιουργήσουν μεγαλύτερη ευημερία για την κοινωνία και του πολίτε. Από το 2010 η υπηρεσία μας έχει επενδύσει περίπου 100 εκατομμύρια για τη δημιουργία δυνατοτήτων σε εθνικό επίπεδο ε, μέσω ενός δικτύου πνευματικής ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε κοινά εργαλεία, κοινέ πρακτικές προς όφελος των χρηστών και η ικανοποίηση των χρηστών έχει αυξηθεί σε αυτό το χρονικό διάστημα. Ε, στην τελευταία μελέτη ικανοποίηση χρηστών Φτάσαμε στο 89% σε σχέση με το 72% ικανοποίηση σε σχέση με πριν από κάποια χρόνια. Ήρθε η στιγμή ε, πλέον αυτό το δίκτυο τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την Πνευματική Ιδιοκτησία να αρχίσει να λειτουργεί, να λειτουργεί για να αντιμετωπίσει τι πιο επίγουσε προτεραιότητε που αντιμετωπίζει το σύστημα πνευματική ιδιοκτησία και να αυξήσουμε έτσι τον αντίκτυπο τη δράση μα. Ε, θέλουμε να συνεισφέρουμε στην ανταγωνιστικότητα, στη δημιουργία ε, θέσεων εργασία ποιοτικών, καλοπληρωμένων υπάρχει ανάγκη να υποστηρίξουμε ιδιαίτερα τι μικρομεσαίες επιχειρήσει που υποχρησιμοποιούν ε, την, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησία. Δείχνουν οι έρευνε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, αποτελούν 99% των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο μία στι 10 από αυτέ όμω έχει οποιαδήποτε μορφή ε, καταγεγραμμένων ε, πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτέ οι εταιρείε όμω που έχουν πνευματικά δικαιώματα καταχωρημένα και προστατευμένα έχουν τι πιθανότητε να μεγαλώσουν και να πετύχουν αυτό είναι και το πλαίσιο του, νέου στρατηγικού σχεδίου μας. Ε, για ένα πολύ σημαντικό έγγραφο στρατηγικού επίπεδου και θα συμπεριληφθεί στο, στο, επίσημο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών. Ε, οι πιο σημαντικές προκλήσεις στα πλαίσια αυτού του στρατηγικού σχεδιασμού είναι να εξασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσουμε να, να προσφέρουμε προσθέμενη αξία σε επίπεδο πνευματική για τι πολίτε και τι επιχειρήσει. Ε, για να πετύχουμε αυτό το όραμα, το σχέδιό μα έχει βασιστεί σε τρει πυλώνε, σε τρει ε, κατευθύνσει, αν θέλετε, ε, για να αλλάξουμε. Είναι εξίσου σημαντική όλοι αυτοί οι τομείς. μία έχει να κάνει του εμπλεκόμενου φορεί, η άλλη έχει να κάνει του πελάτε και η άλλη είναι η εσωτερική, ο εσωτερικό μετασχηματισμό που θα είναι απαραίτητο. Πολύ σύντομα, ε, σε ό,τι αφορά του εμπλεκόμενου φορεί, θέλουμε να δικοποιήσουμε την ευρωπαϊκή συνεργασία για την πνευματική ιδιοκτησία και να έχουμε περισσότερο άμεσο αποτέλεσμα ε, για τι επιχειρήσει. Ε, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τι προχωρημένε πρακτικέ, τα προχωρημένα εργαλεία στα πλαίσια του δικτύου πνευματική ιδιοκτησία του Ευρωπαϊκού. Θα πρέπει να ενισχύσουμε την εφαρμογή, να δημιουργήσουμε ένα hub γνώσεων. Αυτό θα δώσει ένα μεγαλύτερο ρόλο στα κράτη-μέλη και στα γραφεία πνευματική ιδιοκτησία, στα εθνικά, έτσι ώστε να βοηθηθούν οι μικρομεσαίε επιχειρήσει σε επίπεδο εφαρμογής. Αυτό θα υποστηριχθεί μέσω ευρωπαϊκών project που θα προχωρήσουν παράλληλα. Ένα βασικό στόχο είναι να συνεχίσουμε να δημιουργούμε δυνατότητε στα πλαίσια του συστήματο πνευματική διοκτησία, χωρί να υπάρχει όμω επικάλυψη προσπαθειών και αυξάνοντα ε, την εγκύτητα με του χρήστε. Τα εθνικά γραφεία είναι πιο κοντά στι μικρομεσαίε επιχειρήσει ε, στι οποίε θέλουμε να φτάσουμε, μιλούν και τη γλώσσα του, είναι, είναι πιο εύκολο να συντονιστούν σε εθνικό επίπεδο. Το γραφείο έχει διαπιστώσει ότι για να μπορέσει να πετύχει στρατηγική είναι σημαντικό να υπάρξει μια καλή επικοινωνία, να υπάρξει μια συνεργασία και με όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Λαμβάνοντα υπόψη το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διακυβέρνηση του EUIPO, θέλουμε να εμβαθύνουμε την επικοινωνία με το Κοινοβούλιο και τα μέλη του και να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε επίση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε αυτό το πλαίσιο θέλω να σα ευχαριστήσω για τους ορισμούς συμμετοχής ε, ε, στο παρατηρητήριο και βεβαίως θα συνεργαστούμε στενά με τα μέλη τα οποία θα ορίσετε για να συμμετάσχουν απευθείας στην διακυβέρνηση του γραφείου, στη Διαχειριστική Επιτροπή και στην Επιτροπή Προπολογισμού. Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στις προτεραιότητες που αλλάζουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο των τομέα των ευρωπαϊκών και των σχετικών δικαιωμάτων και το στρατηγικό μα σχέδιο, σχέδιο θα μα βοηθήσει για να πετύχουμε αυτού του στόχου. Είναι ο δικό κατά κάποιο τρόπο. Θα ήθελα τώρα να περάσω στο δεύτερο πυλώνα ε, που έχει να κάνει με τους πελάτες. Ε, και βεβαίως αυτό συνδέεται με το δίκτυο και τα δίκτυα στα οποία αναφερθήκαμε. Πολλές ως πρωτοβουλίες θα προκύψουν από εκεί, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις και οι πολίτες να μπορέσουν να προχωρήσουν. Ιδιαίτερα οι πελάτες ε, του, της υπηρεσίας μας. Με μια πιο διαφοροποιημένη προσέγγιση τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα. Θα επικεντρωθούμε λοιπόν στις ανάγκες της κάθε ομάδας ε, πελατών πιο κατακαιρματισμένα, ε, πιο στοχοθετημένα. Θα έχουμε μια, μια πιο πλήρη υποστήριξη ε, ήδη πριν την υποβολή αίτηση έω και την εφαρμογή. Ιδιαίτερα για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Θα υπάρξει λοιπόν ένα ειδικό πρόγραμμα για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει και θα προτείνουμε τη δημιουργία μια ιστοσελίδα σε 22 γλώσσε που θα συμπληρώνεται με λειτουργίες εχμής. Μιλάμε για chatbots σε 22 γλώσσες, ε, μηχανές αναζήτησης κτλ. Θέλουμε επίσης να διευκολύνουμε την εφαρμογή των δικαιωμάτων IP ε, σε πλατφόρμες ε, ηλεκτρονικού εμπορίου. Το σχέδιό μας θα είναι το όχημα και για πιο φιλόδοξες αλλαγές εφόσον υπάρξει πολιτική και θεσμική βούληση. Παραδείγματο χάρη, μέρος του προγράμματός μας και του των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, είναι ο εξορθολογισμό πολλών πρωτοβουλειών που έχουν ω στόχο τι μικρομεσαίε επιχειρήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω προχωρημένων εργαλείων πληροφορική, help desk, και έτσι μπορούμε να βοηθήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση που θέλει να δημιουργήσει κάποια trust fund ή παρεμφερή εργαλεία χρησιμοποιώντα ε, κάποιο από το πλεόνασμα τη υπηρεσία μα, εφόσον βεβαίω αυτό εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με πρωτοβουλίε των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, έχει να κάνει και με την εφαρμογή ε, προγραμμάτων που χρηματοδοτούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να υπάρξουν ίσε ευκαιρίε ε, σε τομεί προτεραιότητα στην Κίνα, στην Αφρική, προ όφελο των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Αναφέρθηκα λοιπόν στους δύο πυλώνες του σχεδίου μας, ε, μπλεκόμενοι φορείς και πελάτες. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα στοιχεία, αλλά διαπιστώσαμε ότι η τεχνολογία αλλάζει και επηρεάζει, καθορίζει το τι μπορούμε και τι πρέπει να κάνουμε, θα πρέπει να έχουμε και άριστους υπαλλήλους. Έτσι λοιπόν το τρίτος ε, στόχος μας, ο τρίτος πυλώνας είναι πιο πολύ εσωτερικός Αναγνωρίζουμε δηλαδή ότι επειδή έχει επιτύχει το σύστημα το χρηματοδότησης της μα, μας, υπάρχει και οικονομική βιωσιμότητα και αυτονομία δηλαδή, είναι σημαντικό από εκεί πέρα να συνεχίσουμε ε, να προσπαθούμε να είμαστε ακόμα πιο διαφανεί και να λογοδοτούμε περισσότερο. Ε, είμαστε αποτελεσματικοί οικονομικά, διότι χρησιμοποιούμε νέα ε, μοντέρνα εργαλεία για τον προγραμματισμό, τις εκθέσεις, τις προμήθειες, όπως και με άλλα project ε, μετασχηματισμού η χρήση τεχνητής νοημοσύνης, data analytics, ε, ίσως να μας βοηθήσει ε, για να έχουμε πιο προχωρημένα συστήματα αναφοράς και ανάλυσης. Θα εξακολουθούμε βεβαίως να τηρούμε τα υψηλότερα πρότυπα εξωτερικού ελέγχου και μέτρων κατά της απάτης για να εξασφαλίσουμε και τους πελάτες μας. Θέλουμε επίσης να αναπτυχθούμε σε επίπεδο δεξιοτήτων, να δώσουμε έμφαση στην διαβίου μάθηση και στη συμμετοχή του προσωπικού. Ε, θέλουμε να ε, εκμεταλλευτούμε την ψηφιακή εποχή Θέλουμε επίσης να είμαστε ακόμα πιο βιώσιμοι, δίνοντας έμφαση στη μείωση των αποβλήτων νέων τεχνολογιών, οι οποίες θα, θα πληρούν τα περιβαλλοντικά πρότυπα. Θέλουμε να μειώσουμε το αποτύπωμα άνθρακα, ε, μέτρα που έχουν ως στόχο μείωση των εκπομπών ε, αερίων του θερμοκηπίου επίσης ε, θα παρθούν. Πρόκειται για σημαντικές προκλήσεις, αλλά σας, σας διαβεβαιώ ότι το προσωπικό μας ε, έχει δείξει στα δύο προηγούμενα σχέδια ότι είμαστε ικανοί να το φέρουμε σε πέρα αυτό, είμαστε διαθέσιμοι, έχουμε τη βούληση και πιστεύω αυτό θα γίνει και στο επόμενο χρονικό διάστημα. Βεβαίω, το χρονοδιάγραμμα για το επόμενο στρατηγικό σχέδιο, μετά και την πρώτη φάση διαβούλευση στο δεύτερο τρίμηνο του εξάμενου, υπευλήθη στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην Επιτροπή Προπολογισμού τον Ιούνιο και, έλαβε, και έτυχε σημαντική στήριξη. Στο στρατηγικό σχέδιο στη συνέχεια προσαρμόστηκε και μια, ένα δεύτερο κύμα δημοσίων διαβουλεύσεων με το νέο αυτό, και για το νέο αυτό σχέδιο έλαβε χώρα έω τα μέσα Σεπτεμβρίου. Μετά από τη συνεισφορά όλων και αυτή τη αλλαγή απόψεων, ε, το τελικό σχέδιο θα υποβληθεί προ έγκριση τον Νοέμβριο στο Διοικητικό Συμβούλιο και θα ξεκινήσει από εκεί και πέρα η εφαρμογή του από τον Ιούλιο του χρόνου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, εκπροσωπείται βεβαίω στο Διοικητικό Συμβούλιο, έχει τη δική του ευθύνη για να συμμετέχει στη διαδικασία λήψη αποφάσεων για αυτό το νέο στρατηγικό σχέδιο. Είναι λοιπόν σημαντικό για την υπηρεσία μα να λάβει την υποστήριξη αυτή τη Επιτροπή εν ώψη τη συνεδρία του Νοεμβρίου. Το επίπεδο φιλοδοξία που περιλαμβάνει το έγγραφο αυτό είναι ήδη ψηλό. Όμω με την υποστήριξη και τη βοήθεια ε, των Ευρωπαϊκών Συμφωνών Οργάνων θα, προχωρήσει ακόμα περισσότερο. Το σχέδιό μα είναι η απαρχή μια σειρά από μέτρων που χρειάζονται θεσμική υποστήριξη για να εφαρμοστούν αποτελεσματικά. Και αυτό θα διευκολυνθεί και από το νομοθετικό έργο. Θα ήθελα να αφαιρθώ σε δύο τομεί προτεραιότητα στα πλαίσια του, του σχεδίου αυτού, όπου υπάρχει ανάγκη μεγαλύτερου συντονισμού έτσι ώστε να βοηθηθούν οι μικρομεσαίε επιχειρήσει και να αντιμετωπίσουμε το θέμα τη ε, εφαρμογή. Για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, αν θέλουμε να τι βοηθήσουμε για να χρησιμοποιήσουν τα πνευματικά δικαιώματα και να τα εκμεταλλευτούν, πρέπει να είναι πιο απλό το τοπίο. Δεν θέλουν οι μικρομεσαίε επιχειρήσει να έχουν να αντιμετωπίσουν πολλέ και διάφορε υπηρεσίε και γραφεία που είναι υπεύθυνα για τι διάφορε μορφέ υποστήριξη ή διάφορα εργαλεία για την πνευματική ιδιοκτησία. Θέλουν ένα ενιαίο συνομιλητή. Ε, θέλουν απλοποιημένη, προσβάσιμη δυνατότητα ε, για την επίλυση των όποιων διαφορών. Αυτό δεν έχει να κάνει με τα σήματα, έχει να κάνει και με το εμπορικό απόρριτο, ε, ε, γεωγραφικές ενδείξεις κλπ. Η EUIPO λοιπόν είναι στην καλύτερη θέση για να είναι αυτός ο ενιαίος συνομιλητής. Αλλά πρέπει να το χωρίσουμε βήμα-βήμα. Εννοείται ότι τα πράγματα θα πάνε πιο γρήγορα με την θεσμική υποστήριξη. Στον τομέα, παραδείγματο χάρη του design, θα συνεχίσουμε επίση να υπάρχει πίεση για την νομοθετική μεταρρύθμιση που εξετάζει ήδη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμεί είμαστε έτοιμοι να συνεισφέρουμε σε αυτό, εφόσον μα ζητηθεί, ε, διότι τα δικαιώματα design είναι εξαιρετικά προσβάσιμα που μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν τι νομικέ επιχειρήσει. Κυρίε και κύριοι, αξιότιμα μέλη τη Επιτροπή, κυρία Πρόεδρε, ε, το 2025 ε, δείχνει την κατεύθυνση, δείχνει το δρόμο. Είναι το πλαίσιο που θα μας κατευθύνει για να πετύχουμε να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προτεραιότητες στον τομέα των πνευματικών ε, δικαιωμάτων να αποκοινούμε με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Τα τελευταία 25 χρόνια η e UIPO σιγά σιγά έχει λάβει μεγαλύτερε ευθύνε στον τομέα των πνευματικών δικαιωμάτων για να αυξηθεί η προσθέμενη αξία του και ο αντίκτυπό του στην ανταγωνιστικότητα και στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και τη κοινωνία γενικότερα. Τα έχουμε κάνει όλα αυτά με μηδενικό κόστο για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Και εφόσον αυτό το μοντέλο αυτοχρηματοδότησης έχει πετύχει. Ε, νομίζω ότι έτσι πρέπει να συνεχίσουμε. Με τη βοήθειά σας και με το απαραίτητο νομοθετικό έργο ε, που θα πρέπει να ακολουθήσει, μπορεί αυτό να επεκταθεί και σε άλλους τομείς προς όφελος των επιχειρήσεων. Θα ήθελα να πω ότι αυτός είναι ο δρόμος ε, και το όχημα για να το πετύχουμε είναι το στρατηγικό μας και ελπίζω να υποστηρίξετε αυτό το όραμα στο μέλλον, όπως και το πράξετε και στο παρελθόν. Τέλος, ε, με βάση τις προθέσεις τη υπηρεσία μα να ενισχύσουμε τι σχέσει με τα θεσμικά όργανα, θα μπορούμε να πάμε και πέρα από αυτή την, την, την επίσημη δηλαδή, απόψε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα και να υποβάλουμε μια επικαιροποίηση, μια ενημέρωση μια φορά το χρόνο στην Επιτροπή σα. Καλό επίση τα μέλη τη επιτροπή, σα, εφόσον θεωρείτε σκόπιμο, να έρθετε να μα επισκεφτείτε, να δείτε πώ εργαζόμαστε, όπου χίλια άτομα προσωπικό και περίπου 500 υποστηρικτικό προσωπικό ε, στο Αλικάντε εργάζονται ακούραστα για να παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητα προς τους χρήστε. Σα ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία αυτή και είμαι έτοιμος να ακούσω τα ερωτήματά σας. Ευχαριστώ. Um, uh, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά που μας είπατε ε, και σχετικά με το στρατηγικό σχεδιασμό σας 2025. Αν θέλουν τα μέλη να πάρουν το λόγο, παρακαλώ κύριε συνάδελφε. Ευχαριστώ πολύ ε, κύριε Πρόεδρε, ε, κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Μια σύντομη ερώτηση ενδεχομένως και στο Executive Summary αλλά και στο προσχέδιο του στρατηγικού σχεδιασμού αναφέρεται ότι η υπηρεσία θα ενδυναμώσει την ε, επαφή με το Κοινοβούλιο και τα μέλη του Κοινοβουλίου θεωρώντας ότι είναι σημαντικός ο ρόλος του Κοινοβουλίου κατά την έννοια αυτή. Επίσης, ε, σαφής... Ε, εγώ θα ενδιαφερόμουν πάντως να μου πείτε ή να καταλάβω εάν προβλέπετε οποιαδήποτε συγκεκριμένη δράση συνέργειας με την Επιτροπή μας εκτός από αυτές τις εθιμοτυπικές ας πούμε επαφές. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση, η πιο σύντομη. Δεύτερη, αναφερθήκατε στον τρίτο πυλώνα στρατηγικής προώθησης, ας πούμε, ε, και αναφερθήκατε σε τις ε, ε, στην καινοτομία, στη, στον τόπο εργασίας ε, και λέτε ότι θα πρέπει με πολύ προσεκτικό τρόπο να αντιμετωπιστεί η μετάβαση της εργασίας στην αυτοματοποίηση, ε, στην υλοποίηση των νέων τεχνολογιών, cloud computing, blockchain κλπ. Αυτές οι ιδέες αναφέρονται άλλωστε και στη σελίδα 5 του προσχεδίου, του στρατηγικού σχεδιασμού, όπου αναφέρεται ότι θα πρέπει να εφαρμοστούν οι νέες τεχνολογίες και σε συνεργασία με τα άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τούτων λεχθέντων. Μήπως θα μπορούσατε να είστε πιο συγκεκριμένος σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ε, θα ε, ε, σχετίσετε αυτές τις τεχνολογίες με τον στρατηγικό σας σχεδιασμό και επίσης μέχρι ποιο βαθμό ε, θα χρησιμοποιήσετε τις ε, διεθνείς, ε, τα διεθνή διδάγματα και σε ποιο βαθμό θα έχετε ως στόχο την ανταλλαγή τέτοιων στοιχείων με άλλους οργανισμούς προστασίας διανοητικής ιδιοκτησίας και πώς θα διασφαλίσετε και την προστασία στρατηγικών πληροφοριών. Ένα άλλο στοιχείο. Υπάρχει μία ε, βασική πρωτοβουλία για την καλύτερη κατανόηση της διανοητικής ιδιοκτησίας και περιλαμβάνει ε, από εκστρατείες ευαισθητοποίησης μέχρι συγκεκριμένα ε, προγράμματα. Όλα αυτά εμείς ως σοσιαλιστές και δημοκράτες τα καλωσορίζουμε γιατί με τον τρόπο αυτό μπορεί ο μέσος Ευρωπαίος πολίτης να διευρύνει τη γνώση του σχετικά με το τι σημαίνει διανοητική ιδιοκτησία. Ιδιαιτέρως το προσχέδιο του στρατηγικού σχεδιασμού αναφέρει ότι θα υπάρξουν δράσεις ε, έτσι ώστε οι πολίτες να μπορούν να καταλάβουν ποια είναι ε, προϊόντα ε, πλαστά, απομίμησης ή που δεν φέρουν το σωστό εμπορικό σήμα, το αυθεντικό εμπορικό σήμα. Ευχαριστώ. Απάντηση. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Πρώτον, ε, όσον αφορά την ανταλλαγή απόψεων και την ενίσχυση της συνεργασίας με την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Ε, είπα και στην αρχική μου ομιλία ότι προτίθεμαι να ξεπεράσω την ε, εθνική παρουσίαση αναπενταετία των στόχων. Το αναφέρω αυτό γιατί θέλω πραγματικά μία φορά το χρόνο να κάνω τη σχετική αναφορά δράσεων και δραστηριοτήτων στην, Ευρωπαϊ... στην δική σας Επιτροπή σε σχέση και με το στρατηγικό σχεδιασμό. Όπως είπα και προηγουμένως, θα καλέσουμε όλα τα μέλη της Επιτροπής σας να μας επισκεφθείτε στο Αλικάντε και βεβαίως θα εργαστούμε ε, στενά με οποιοδήποτε εκπρόσωπο ορίσετε ε, στο ε, διοικητικό ε, συμβούλιο ε, ή στο παρατηρητήριο. Στα πλαίσια δε αυτού του παρατηρητηρίου θα έχουμε ευρέω την δυνατότητα να ανταλλάξουμε απόψεις και ιδέες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να βοηθήσουμε και τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Δεύτερη ερώτηση όσον αφορά την ε, τροποποίηση, την μεταρρύθμιση της ε, υπηρεσίας. Θέλουμε ε, να χρησιμοποιήσουμε σωστά τις νέες τεχνολογίες, λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο που η χρήση τους θα έχει στο εργατικό δυναμικό. Θέλουμε να υλοποιήσουμε την μετάβαση αυτή με πολλούς τρόπους. Πρώτα απ' όλα, Έχουμε ε, καταβάλει μεγάλες προσπάθειες τα τελευταία χρόνια για την αυτοποίηση ε, της ε, καταγραφής των εμπορικών σημάτων και του σχεδιασμού design. Τώρα θέλουμε όμως να δώσουμε μια νέα όθηση στην καταγραφή μεσολογισμικού αυτού της, ε, της διαδικασίας. Ε, βεβαίως έχουμε τη δέσμευση των γλωσσών γιατί δουλεύουμε με 23 ε, γλώσσες Δουλεύουμε επίσης με διαδικασίες machine learning, καθώς επίσης και πρόσβαση σε αυτοματοποιημένη μετάφραση, έτσι ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική η εργασία, μου, η εργασία μας. Αυτό σημαίνει ότι κάποια από τα προφίλ και τις δεξιότητες του προσωπικού θα πρέπει να αλλάξει, γιατί κάποιες θέσεις θα καλυφθούν από την αυτοματοποίηση, αλλά βεβαίως η εργασία ε, και το εύρος εργασιών της υπηρεσίας μας διευρύνεται άρα θέλουμε προσωπικό που να ανταποκρίνεται στις νέες λειτουργίες μας. Ε, εάν θέλει κανείς να εφαρμόσει την data analytics ή την ε, διανοητική ε, την artificial intelligence ε, ή οτιδήποτε ε, παρόμοιο, ε, αυτό που θέλουμε στην ουσία είναι να είμαστε ανταγωνιστικοί και να μπορούμε να προσφέρουμε αυτά που ζητά η πλευρά της ζήτησης. Γι' αυτό λοιπόν ξεκινάμε συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα έτσι ώστε φοιτητέ να μας βοηθήσουν στην χρήση νέων τεχνολογιών και την μελέτη των νέων τεχνολογιών η ισορροπία πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει όσον αφορά την μετάβαση των εργαζομένων και στην απόκτηση αυτών των νέων ε, δεξιοτήτων. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ε, ε, κυρίως να διατηρήσουμε τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα. Η τρίτη σας ερώτηση όσον αφορά την καλύτερη κατανόηση των, της έννοιας της διανοητικής ιδιοκτησίας. Έχουμε αρκετές ε, πρωτοβουλίες ε, σχεδιάσει ήδη. Ε, μας ρωτήσατε, ας πούμε, ε, να δώσουμε κάποια παραδείγματα δραστηριοτήτων που μπορούν να βοηθήσουν τους ε, πολίτες να καταλαβαίνουν τη διαφορά ανάμεσα στο παράνομο ε, περιεχόμενο και το νόμιμο ή τα fake προϊόντα, τα πλαστά προϊόντα. Κοιτάξτε, ένας από τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε στην μείωση στην ουσία, την πρόσβαση αυτών των παράνομων προϊόντων είναι να αυξήσουμε την νόμιμη προσφορά. Το κάνουμε αυτό όσον αφορά το copyright με το πρόγραμμα Αγκορατέκα. Επίσης, θέλουμε να ε, δημιουργήσουμε ε, μία βάση ε, προσβάσιμη από το Offenwork. Επίσης, μια βάση ε, δεδομένων μέχρι τον Ιούνιο του 2021, που θα αντιλεί στοιχεία από την αγορά και το εμπόριο. Γενικά, πάντως, θέλουμε, προτιθέμεθα να συνεχίσουμε να τροφοδοτούμε τη συζήτηση σχετικά με παραβιάσεις ε, γενικότερες, αλλά ε, ε, κυρίως όσον αφορά τα πλαστά προϊόντα και τα θέματα ασφαλείας. Δεν αναφέρομαι μονάχα σε φάρμακα. Πρόσφατα, ας πούμε, μαζί με την Europol καταφέραμε να σταματήσουμε μια εγκληματική συμμορία η οποία ε, βιομηχανικό γάλα σε σκόνη ε, το ξανασυσκεύαζε έτσι ώστε ε, να είναι γάλα για βρέφη σε σκόνη και έχουμε και ευρύ πρόγραμμα συνεργασίας με την ε, Europol και άλλες ε, διεθνείς αρχές επιβολής δικαίου ε, και σιγά σιγά κερδίζουμε και έδαφος και όσον αφορά τα θέματα αυτά. Αυτά νομίζω για την ώρα όσον αφορά αυτές τις ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πολύ για τις ερωτήσεις Μια άλλη ερώτηση παρακαλώ. Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση. Θα Κάνω και εγώ την ερώτησή μου. Λοιπόν, σα ευχαριστώ που μα ενημερώσετε για τι ε, νέε προκλήσει του στρατηγικού σχεδίου του γραφείου και είναι σημαντικό να παίξουν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ένα ρόλο εκεί πέρα. Αναφέρατε την αξία της πνευματικής ιδιοκτησίας η οποία αυξάνεται αλλά ταυτόχρονα οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις έχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα με την δήλωση και διασφάλιση της πνευματικής ιδιοκτησίας τους. Οπότε είναι σημαντικό να δούμε και το τι, πώς θα επηρεάσει η τεχνητή νοημοσύνη το θέμα αυτό. Οπότε αυτό το οποίο θα με ενδιαφέρει είναι πότε σκοπεύετε ακριβώς να δείτε τις δυνατότητες ε, και το πώς θα επηρεάσει η τεχνητή νοημοσύνη το θέμα αυτό και αν μπορείτε να στηρίξετε τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Και το ερώτημα του εάν ε, ειδικά στο θέμα της παραποίησης προϊόντων ή διασφάλισης της ποιότητας ε, των προϊόντων υπάρχουν κάποια αποτελέσματα ή αν πρέπει να καταλήξουμε σε κάποια άλλα μέσα με βάση τις εμπειρίες που έχετε σε συνεργασία με την ε, Europol. Αυτά και σας ευχαριστώ για την ε, συνεργασία με την Επιτροπή μας. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, όταν κοιτάμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Ήδη έχουμε μία ιδέα με βάση τις μελέτες που έχουμε κάνει για το ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, τα βασικότερα είναι ότι δεν είναι ακόμα αντιληπτά τα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και η αξία τους από τις ε, εταιρείε αυτές. Προσφάτως κάναμε κάποιες ε, συνεντεύξεις με 8.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι μισές είχαν πνευματικά δικαιώματα, οι άλλες μισές όχι. Για να δούμε για ποιους λόγους ε, έκαναν κάποια εγγραφή και αν δεν είχαν κάνει τι θα χρειαζόταν για να τους προσελκύσει το σύστημα για αυτούς που είχαν κάνει εγγραφή. Ένα, στο, ένα 60% θεώρησαν ότι ήταν χρήσιμο για να αποτρέψουν παραβίαση των δικαιωμάτων τους ε, αντιγραφή και κλοπή μυστικών. Επίσης αναφέρθηκε η νομική βεβαιότητα και το θετικό αποτέλεσμα στην εικόνα της εταιρεία. Για αυτές που δεν είχαν καταθέσει κάποιο δίπλωμα, είναι ότι δεν υπάρχει κάποια γνώση για το πώς λειτουργεί το σύστημα αυτό και μετά υπάρχει το θέμα του κόστους της προσφυγής στα δικαστήρια, όχι τόσο της καταγραφής γιατί με 950 ευρώ μπορεί να κατοχυρωθεί ένα εμπορικό σήμα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα μονοπόλιο για 10 έτη. Οπότε νομίζω αξίζει. Αλλά βεβαίως η επιβολή αυτών των δικαιωμάτων σε περίπτωση παραβίασης και βεβαίως ε, οι καυγάδες στους οποίους μπορείς να μπλέξεις κατά τη διάρκεια της ε, καταγραφής από εταιρείε ε, που αντιτίθενται είναι τα προβλήματα που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε. Οπότε, πώς σκοπεύουμε να τα, αντιμετωπίσουμε. Από την ε, σκοπιά των πληροφοριών θεωρώ ότι έχουμε πέσει θύμα της υπερβολικής πληροφόρησης που πλέον ε, δεν έχει σωστή δομή, δηλαδή εντός ε, του θεσμικού οργάνου μας για την ε, έντολη μας έχουμε δει πάνω από 800 ε, πρωτοβουλίες με links στο σελίδες που άλλα δεν ισχύουν. Οπότε μια πρώτη χαρτογράφηση του τι υπάρχει, τι εξακολουθεί να ισχύει και πώς μπορούμε να απλοποιήσουμε αυτό το τοπίο σε κάποιες πληροφορίες που θα είναι εύκολα κατανοητές είναι μεγάλο κομμάτι της δουλειά μας. Μετά, όταν έχουμε αυτές τις πληροφορίες πρέπει να τις ε, διαδώσουμε. Δηλαδή, με site, με chatbot, με αυτόματη μετάφραση, αλλά όπως είπα ε, πρέπει και εμείς να συνεργαστούμε με τις εθνικές υπερορίες και μπορούμε έτσι να χρηματοδοτήσουμε κάποιες εθνικές δραστηριότητες για να προσελκύσουμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και αυτό δεν θα γίνει με το να τις φέρουμε σε ένα συνέδριο στην Εθνική Υπηρεσία. Πρέπει να πάμε στα εμπορικά επιμελητήρια, στην Ένωση των Συμβολογράφων και τα σχετικά, για να ενημερωθούν για αυτά τα ζητήματα. Μετά, εάν αποφασίσουν να καταγράψουν κάτι, θέλουμε να δούμε το θέμα των διαφωνιών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ε, καταγραφής με το να προωθήσουμε την ε, εναλλακτική επίλυση διαφορών. Οπότε η άτυπη, αν θέλετε, διαμεσολάβηση είναι κάτι το οποίο μπορούμε να δούμε. Μπορούμε βέβαια να πάμε και στην διαιτησία, γιατί οι διαφωνίες δεν αφορούν μόνο τα εμπορικά σήματα, αλλά διευθύνσει διαδικτύου ή ονόματα εταιριών και εκεί πέρα δεν έχουμε κάποια αρμοδιότητα. Άλλα γραφεία πνευματικής ιδιοκτησίας έχουν, εμείς όχι. Οπότε αυτό το οποίο θα θέλαμε εμείς είναι να προσεγγίσουμε διάφορους ενδιάμεσους που παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες και με βάση μια χάρτα να μπορέσουμε να τους προτείνουμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να υπάρχει ένα μητρό, αν θέλετε, του που μπορεί να απευθυνθεί κανείς στην περίπτωση που αντιμετωπίσει προβλήματα. Και μετά, στην επιβολή, και εκεί πέρα θέλουμε ακριβώς να δούμε την επαφή με τα εθνικά γραφεία. Έχουμε συνεργασία με πολλές άλλες ε, υπηρεσίες και έχουμε έτσι καταφέρει να γίνουμε ένας de facto συντονιστής ε, της μάχης ε, κατά της παραβίασης των σημάτων αυτών. Συνεργαζόμαστε με τη ΣΕΠΟΛ, την Europol, τη Γενική Διεύθυνση Ταξούντ της Κομισιόν. Έχουμε διάφορους δηλαδή φορείς που συντονίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οπότε όταν πάμε στο ευρωπαϊκό επίπεδο ε, για να επιβληθούν αυτά τα δικαιώματα πρέπει να πάει κανείς ε, στον δικαστή, έναν εισαγγελέα που δεν αντιλαμβάνεται τα θέματα αυτά, δεν ε, συνειδητοποιεί πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα και νομίζω ότι εκεί πέρα υπάρχει ένας ρόλος που μπορούν να παίξουν οι εθνικές υπηρεσίες για να γίνουν οι εθνικοί συντονιστές είτε έχουν αρμοδιότητα είτε όχι. Νομίζω πως είναι θέμα πληροφόρησης, ε, εκπαίδευσης και συνεργαζόμαστε πολύ με την Ευρωπαϊκή Σχολή Αστυνομίας και Βεβαίω, ε, αυτά είναι και στην διάθεση των εθνικών υπηρεσιών. Οπότε έχουμε αυτό, έχουμε τις ε, εθνικές Βάσει δεδομένων και θεωρούμε ότι μπορούμε να βελτιώσουμε την μάχη που δίνουμε υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριος Φως. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να σας ευχαριστήσω για αυτά τα οποία μας ε, είπατε. Απαντήσατε πολλά πράγματα που ήθελα να ρωτήσω. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω έτσι όπως μας τα παρουσιάσατε αυτά τα σχέδια να συνεχίσετε έτσι με αυτήν την φιλοδοξία. Βεβαίως είναι αυτό το οποίο είπαν οι συνάδελφοι. Η εκστρατεία ευαισθητοποίησης είναι κάτι στο οποίο πρέπει να δοθεί περισσότερο βάρος ε, όταν έχουμε αυτήν την παγκόσμια επαφή και σχέση με την ε, πνευματική ιδιοκτησία που είναι κάτι το οποίο έχουμε αμελήσει και είναι κάτι το οποίο πρέπει να ενισχυθεί, να έχουμε πιο γρήγορες ε, διαδικασίες και απλοποιημένες όταν μιλάμε για τον ψηφιακό τομέα ή οτιδήποτε άλλο και με χρήση αλγορίθμων ή ε, οτιδήποτε χρειάζεται. Ε, για τις κυρώσεις μιλήσατε για συγκεκριμένες ε, νομοθετικές πτυχές. Νομίζω πως όλοι είμαστε ανοιχτοί όταν μιλάμε για επίλυση διαφορών, ειδικά όταν αυτό γίνεται χωρίς αλλαγή του προϋπολογισμού, οπωσδήποτε θα μας βοηθήσει γιατί γενικώ έχω την αίσθηση ότι οι διαδικασίες μας εντωμεταξύ διαρκούν πάρα πολύ. Οπότε θα μπορούσε να προχωρήσει εκεί η διαμεσολάβηση. Το στρατηγικά σχέδια ε, μια φορά το χρόνο ναι. θα πρέπει όμως να είμαστε και φιλόδοξοι Και βεβαίως χρειαζόμαστε νέες απαντήσεις, ε, νέες λύσεις. αυτό θα μας ε, βοηθούσε πάρα πολύ. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναφέρθηκαν ήδη κάποια πράγματα. Σε ποιο βαθμό δηλαδή μπορεί να υπάρξει κάποια εσωτερική βελτιστοποίηση. Σε όλα αυτά λοιπόν θα ήθελα να σας παρακαλέσω να συνεχίσετε να είστε φιλόδοξοι. Αλλά βεβαίως ε, νομοθετικές αλλαγές, οι επιπρόσθετες υπηρεσίες. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να δούμε κάτι τέτοιο, αλλά βεβαίως ε, χρειάζονται και ανάλογες ε, διατάξεις και μια συνεννόηση με την Κομισιόν οπωσδήποτε. Πήγε όσο πιο γρήγορα βέβαια τόσο το καλύτερο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Βόσε. Ναι, Βεβαίω, είμαστε και θα είμαστε και στο μέλλον φιλόδοξοι. Αυτό ε, σα διαβεβαιώ ότι θα υπάρχει και θα προσπαθούμε πάντα να βρίσκουμε ε, ε, τρόπους έτσι ώστε να μην προσέχουμε πάντα στην δικαιοσύνη όσον αφορά την επίλυση διαφορών. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για μας. Όσον αφορά την τεχνολογία που θα βρίσκεται στο επίκεντρο των προσπαθειών μα τα επόμενα πέντε χρόνια, ε, βλέπουμε, προστρέχουμε στην τεχνολογία με διάφορους τρόπους. Πρώτον μέσα από διεθνείς ε, συνεργασίες. Ε, όλοι βεβαίως ε, μιλάνε για τις νέες τεχνολογίες και για τεχνική, τεχνητή νοημοσύνη, αλλά κανείς δεν ξέρει ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Εμείς θα είμαστε δημιουργικοί. δηλαδή θα δημιουργήσουμε ένα δίκτυο ανθρώπων που ασχολούνται με τα πνευματικά δικαιώματα, έτσι ώστε να δούμε τι σημαίνουν οι νέες τεχνολογίες για μας, ε, πώς μπορούν να μας ε, βοηθήσουν οι τεχνολογίες, γιατί εμείς δεν έχουμε το μονοπόλιο των ιδεών και των λύσεων και να δούμε επίσης εάν υπάρχουν τρόποι ε, να ενδυναμώσουμε τη συνεργασία με άλλες αντίστοιχες υπηρεσίες έτσι ώστε να τρέξουμε κοινά προγράμματα. Δεύτερον, είναι ε, η επικέντρωσή μας στην επιβολή μέσω και του παρατηρητηρίου γιατί θέλουμε να είμαστε αρρωγή ε, μέσω της τεχνολογίας προς τις αρχές επιβολής ε, του νόμου, ας πούμε, και πέρσι δώσαμε δυνατότητα παρακολούθησης ε, της, ε, του προϊόντος από τη δημιουργία του, τη μεταφορά του, την, ε, το τελωνείο, την διεμπόρευση, τον, τον χονδρέμπορο, τον λιανέμπορο, τον δεύτερο λιανέμπορο που ενδεχομένως θα ασχοληθεί με την πρόθεση και εμπορία του προϊόντος. Σε αυτήν την διαδικασία blockchain εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε και έχουμε ενημερώσει σχετικά την Επιτροπή τη διαδικασία track and trace που ακριβώς θα ελέγχει το προϊόν σε όλη τη διάρκεια ε, της ε, αλυσίδας. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Ένα άλλο παράδειγμα που έχουμε είναι ένα ε, μητρό IP όσον αφορά την blockchain. Ε, πρέπει να είμαστε σίγουροι βέβαια ότι τα στοιχεία τα οποία βρίσκονται εκεί ε, παραμένουν ε, ακέραια και δεν αναφέρομαι εδώ μονάχα σε δυνατότητα και ενδεχόμενο hacking. Αυτό όσον αφορά την επιβολή του νόμου και εσωτερικά όπως και σας είπα και προηγουμένως, εμείς ξεκινήσαμε ήδη επαφή με ε, ακαδημαϊκά ε, ε, με πανεπιστήμια και τον ακαδημαϊκό κόσμο που ασχολείται με τους υπολογιστές και τα λογισμικά κλπ. έτσι ώστε να έχουμε μια καλή συνεργασία μαζί τους και έτσι ώστε ε, να εξασφαλίσουμε ε, καλή συνεργασία ε, για να μην χρειάζεται να χρησιμοποιούμε και τον προϋπολογισμό που έχουμε για τους μισθούς διότι έχουμε έναν, μια σαφή διαρκή αύξηση του μισθολογικού κόστους μας 3 με 5% κάθε χρόνο και αν δεν βρούμε κάποια λύση θα έχουμε πρόβλημα. Ε, κάποια στιγμή. Επίσης ε, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις σχετικά ε, με αυτοματοποιημένο drafting tool Επίσης, αυτοματοποιημένη μετάφραση ενδεχομένως κάποιων εγγράφων, κάποιων δικαστικών αποφάσεων κλπ. Εμείς 30 εκατομμύρια το χρόνο επενδύουμε ε, στην, ε, σε IT και 2,5 εκατομμύρια αφορούν μονάχα την ε, κυβερνοασφάλεια, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ και μία σύντομη ερώτηση από μένα. Για τους δεσμούς σας με τα πανεπιστήμια και σε ό,τι αφορά την βελτίωση των δεξιοτήτων του προσωπικού σας και για να βοηθήσει τους φοιτητές να βρουν διεξόδους Έχετε λοιπόν σχέσεις με, τις, ε, με τα πανεπιστήμια σε ό,τι αφορά τη συνδρομή που θα μπορούσαν να σας ε, φέρουν για να περάσει το μήνυμά σας προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τα πνευματικά δικαιώματα. Συχνά τα οι εθνικές υπηρεσίες είναι πολύ καλές, αλλά είναι ε, μεγάλες δομέ παρόλα αυτά για μια μικρομεσαία επιχείρηση, η επιχείρηση στο πανεπιστήμιο να είναι πιο, πιο καλός διάβλος. Ναι, βεβαίω. ε, και το κάνουμε. Επειδή το πρόγραμμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, είναι πολύ μεγάλο εν δυνάμει, ε, δεν μπορούμε να αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε όλα αυτά ταυτόχρονα. Κάτι που θα κάνουμε λοιπόν στην αρχή είναι να εντοπίσουμε από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύο-τρεις τομείς τεχνολογίας όπου δραστηριοποιούνται οι α, μικρομεσαίες επιχειρήσεις για ζητήματα πραγματικών δικαιωμάτων και δεν πρόκειται βεβαίω να αντιμετωπίσουμε τις 27 χώρες ε, με μιας. Θα ξεκινήσουμε με δύο-τρεις χώρες, κάποια πιλωτικά προγράμματα, να δούμε αν λειτουργούν και από εκεί και πέρα θα τα διευρύνουμε. Εάν δεν λειτουργήσουν θα τα εγκαταλείψουμε και θα κάνουμε κάτι άλλο. Και βεβαίως τα πανεπιστήμια στους τομέες υψηλής τεχνολογίας όπου έχουμε όλες αυτές τις spin-off ε, ε, είναι σίγουρα ένα εργαλείο που θα χρησιμοποιήσουμε. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βόσης έχει και άλλο ερώτημα. Παρακαλώ. Δεν ξέρω αν το αναφέρατε γιατί ήρθα λίγο αν υπάρξει Brexit. ποιε θα είναι οι επιδράσει ε, και στον δικό σας οργανισμό. Well, I'll call it the million euro question. Ε, είναι η ερώτηση ενό εκατομμυρίου ευρώ, έτσι. Ακούστε, εμείς ε, παρακολουθούμε και ακολουθούμε το άρθρο 50 και τις γραμμές της Κομισιόν. Ε, είμαστε έτοιμοι ε, βεβαίως και για ένα σκληρό Brexit ε, το οποίο θα έχει μεγάλο αντίκτυπο και σε επίπεδο βάσης δεδομένων, συνδέσεις που θα πρέπει να γίνουν, δικαιώματα που θα πρέπει να χωριστούν μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και της υπόλοιπης Ευρώπης, ε, δικαιώματα που υπάρχουν ήδη, αλλά και όλα τα, με, όλες τις διατάξεις, όλες, επιπτώσει, όλα τα σενάρια. Είμαστε έτοιμοι πάντως. Έχουμε τα διάφορα σενάρια, έχουμε τα εργαλεία στη διάθεσή μας. Οποιαδήποτε μορφή συμφωνίας ε, ε που θα οδηγήσει σε βελτίωση ε, σημαίνει ότι δεν χρειαστεί να πάρουμε κάποια από αυτά τα μέτρα. Σε επίπεδο επιχειρήσεων έχουμε δει μετά το δημοψήφισμα μία μείωση στις αιτήσει ε, από εταιρείε ε, ε, που βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, 15% περίπου. Διαπιστώνουμε πάντως ότι υπάρχει μια αλλαγή στο μηχανισμό προστασίας. Κάποιες εταιρείες που στο παρελθόν ε, σε εμάς και το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τώρα περνούν από το άλλο σύστημα προστασίας ε, εμφανίζονται δηλαδή σε εμά μετά, σε δεύτερο, δεύτερο χρόνο. Από πλευρά επιχειρήσεων δηλαδή ο αντίκτυπο είναι περιορισμένο. Σε επιχειρησιακό επίπεδο από την άλλη είμαστε έτοιμοι, είμαστε προετοιμασμένοι ε, για οποιοδήποτε σενάριο. Ευχαριστώ πολύ. Άλλες ερωτήσει. Θα μπορούσα και εγώ να ρωτάω ερωτήσει. να θέλω ερωτήσεις όλη μέρα για τον Brexit, αλλά δεν θα το κάνω. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ε, εντελεχείς εξηγήσεις, πολύ χρήσιμη ενταλλαγή απόψεων. Σας ευχαριστώ κυρία Σαμπό και ε, ανυπομονούμε να συνεργαστούμε και στο μέλλον, στενά. Και τώρα θα περάσουμε στο σημείο 4 της μέσης διάταξης αφορά τις ε, διασυνοριακές ε, συγχωνεύσεις, μετατροπές και ε, αποσχήσεις. Εξετάζουμε το διευθυντικό κείμενο. Σε ό,τι αφορά την οδηγία για whistleblowers και τις γεωγραφικές ενδείξεις, ο φάκελος αυτός υπευλήθη σε ολοκλήρωση μετά την έγκριση Εμεί η Επιτροπή Τζούρι, σύμφωνα με τον κανονισμό 231, θα εξετάσουμε το τελικό κείμενο και θα υποβληθεί στην Ολομέλεια. Αν είμαστε ικανοποιημένοι με το κείμενο, θα το υποβάλουμε ε, προ νομοθετικέ πράξει. Βεβαίω, το εκτιμώντα 31 έχει επανέλθει το κείμενο μετά από πολιτική συμφωνία. Ελπίζω να μην υπάρχει αντίρρηση, μια και η πολιτική συμφωνία είναι αυτό που εγκρίθηκε από την Ολομέλεια. Ε, μπορούμε να υποβάλουμε λοιπόν αυτό το διορθωτικό στην Ολομέλεια. Δεν βλέπω να υπάρχουν αντιρρήσεις. Πολύ ωραία. Σημείο 5. Εφαρμοστικές πράξεις. Ε, δεν υπάρχει κάτι σήμερα. Σημείο 6. Ε, και κλεισμένο το θυρών όμως. Δύο λεπτά διάλειμμα για να προετοιμάσουμε και το web streaming.